Πρόεδρος, συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Περνάμε στην έκθεση Γκρέσλε. Περνάμε λοιπόν στην έκθεση Γκρέσλε. Μία ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Και Πρέπει να δώσω προηγουμένω ε, το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ως Πρόεδρος της Επιτροπής μου ζητήθηκε Δυστυχώς κλείνει το μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, λέει, διάφοροι συνάδελφοι, μέλη της Επιτροπής, μου είπαν ότι έλαβαν γραπτή ενημέρωση από το Γενικό Διευθυντή της Όλαφ για την ε, νομοθετική απόφαση. Εμείς δεν την πήραμε αυτή την ε, ενημέρωση από την ΚΟΝΤ. Δεν είναι σοβαρός τρόπος αυτός αντιμετώπιση του Κοινοβουλίου από έναν επίσημο ευρωπαϊκό θεσμό. Και καλό τον Πρόεδρο να ε, ε, εξετάσει περαιτέρω και να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, λέει ο Πρόεδρος. Θα το λάβω υπόψη μου. Να ψηφίσουμε την έκθεση Γκρέσλε ονομαστική. Άρχεται. Die Πέρας. Η έκθεση δεν συγκέντρωσε την αναγκαία πλειοψηφία. Η κοινή θέση του Συμβουλίου η μη τροποποιηθήσα κοινή θέση του Συμβουλίου θεωρείται λοιπόν ότι ενεκρίθη. Περάμε στο επόμενο θέμα της μέρης διάταξης, έκθεση Giegold. Για την τροπολογία 1 έχει ζητηθεί ψηφοφορία κατά δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές όχι μόνο για το δεύτερο τμήμα έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία τώρα είμαστε στο πρώτο τμήμα για το πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστική άρχεται Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 σε μπε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στο Χ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στο κείμενο της Επιτροπής ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 ΣΕ σε B. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην ψήφιση της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή τώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω αναβολή της τελικής ψηφοφορίας και επαναφορά, αναπομπή δηλαδή στην Επιτροπή, προκειμένου να ξαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο από τη στιγμή που κάνει το Συμβούλιο αυτό που υποχρεούται και να κυρίως να λάβει μια θέση. Ωραία, ψηφίζουμε αυτή την πρόταση του συζητή. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην έκθεση Γκρότε. Τροπολογίες 22, 25 και 27. Όλες μαζί ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτονται. Τροπολογία 21. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε θα ψηφίσουμε τώρα την τροποποιημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. να δώσω τον λόγο στον κύριο εισηγητή. Κύριε Πρόεδρε, με βάση το άρθρο 57 παράγραφος 2 όπως και προηγουμένως θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα να αναβάλουμε την τελική ψηφοφορία επί του νομοθετικού ψηφίσματος για να αναλάβουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ποιος είναι υπέρ αυτής της πρότασης? Κατά Αποχές. Πρέπει να το ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία που ενεκρίθη. Περνάμε στην έκθεση Παγνιού. Τροπολογία 49, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει το μπλοκ 2 Περνάμε στην τροποποιηθήσα πρόταση της Επιτροπής Ονομαστική Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και ε, συγχαρητήρια ε, στον εισηγητή. Περνάμε στην έκθεση υποδηματά για, τις, ε, για το φόρο επί των δημοσιοχρηματοπιστωτικών συναλλαγών συνολικά 1 έως 32, 35 με 38 και 41 έως 54 όλες μαζί ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Για την τροπολογία 33 της Επιτροπής ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 κατά τμήματα ονομαστικές Τμήμα 1. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 ονομαστική άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τώρα λοιπόν Περνάμε στην τροπολογία 56 και 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Ψηφίζουμε το κείμενο της Επιτροπής υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροποποιηθήσα πρόταση Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία επί του νομοθετικού ψηφίσματος άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία και ε, θερμά χαρητήρια στην εισηγήτρια. Περνάμε τώρα στην έκθεση Balts. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, να αξιοποιήσω την ευκαιρία να εκφράσω την απορία μου γιατί για αυτό το σημαντικό θέμα της ε, εισαγωγής του ευρώ στη Λετωνία δεν έγινε καμία συζήτηση αυτή την ομάδα στην Ολομέλεια. Μια σαφής ε, πλειοψηφία στην Επιτροπή δεν σημαίνει πως αυτό το θέμα πρέπει να περνάει στα γρήγορα και με απογοητεύει ιδιαίτερα το ότι η διάσκεψη των Προέδρων απέρριψε το αίτημα της ομάδας μας να γίνει συζήτηση. Είναι σαφής ε, ο λόγος. Δεν θα μπορούσα να ε, θεωρήσω κανένα άλλο θέμα τόσο σημαντικό στην ημερήσια μας διάταξη αυτής της εβδομάδας. Είναι λυπηρό λοιπόν ότι η ένταξη στην Ευρωζώνη της Λετωνίας δεν συζητείται καθόλου. Νομίζω ότι είναι φυσικά ευπρόσδεκτη αυτή η ε, ένταξη και πρέπει να τονίσουμε και τις προσπάθειες που έκανε η χώρα αυτή τα τελευταία χρόνια. Χαίρομαι λοιπόν που η Λετωνία θα μπορέσει, ελπίζω, να ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου του 2014 και πιστεύω ότι έπρεπε να υποθεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, συνάδελφε Μπάλτς. Να περάσουμε στην προφορία. Τροπολογία ένα ονομαστική άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Επίσης ονομαστική άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Επίσης έχει ζητηθεί ονομαστική άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται με ευρύτατη πλειοψηφία θερμά συγχαρητήρια στην Λετωνία. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα για την οδική ασφάλεια. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτω. Ε, εντάξει, άμα θέλετε, ας το ελέγξουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Θα σας παρακαλούσα θερμά να σηκώνετε επαρκώς και επαρκής το χέρι σας. Τροπολογία 1, ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε συνολικά το κείμενο υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα να περάσουμε την έκθεση Ταβάρες. Τροπολογία 1 είναι το εναλλακτικό ψήφισμα μιας πολιτικής ομάδας. Ποιοι είναι υπέρ αυτού του ψηφίσματος. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα. Στις τροπολογίες 2 έως 6 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ να ελέγξουμε. Άρχεται. πέρασε, Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. 69 του αρχικού κειμένου. Δύο τμήματα. Και είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καλώς, να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 70. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 73. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 77 παράγραφος. Επίσης ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 78 ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 79. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 80. Κατά τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 81. Ονομαστική άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. Παράγραφος 85. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε ψηφίζουμε το τροποποιηθέν συνολικό κείμενο ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές εγκρίνεται καλά άμα θέλετε να ελέγξουμε Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε το κοινό ψήφισμα για τις πρόσφατες ε, πλημμύρες στην Ευρώπη. Να ψηφίσουμε το κοινό κείμενο ε, διαφόρων πολιτικών ομάδων. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση Μακάτι. για την ε, διαφορετική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη. Ψηφίζουμε την παράγραφο 4, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9 του αρχικού κειμένου. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, επίσης ονομαστική, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9, εδάφια 2 σε 6 ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνονται. Παράγραφος 9 εδάφιο 7 ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνονται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. Παράγραφος 10. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 13, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική άρχεται. Πέρας. Επίση εγκρίνεται παράγραφος 14 του αρχικού κειμένου. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική άρχεται. Πέρασμα Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την παράγραφο 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Μετά την παράγραφο 16. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 30. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 ονομαστική άρχεται πέρας εγκρίνεται Η αιτιολογική σκέψη ή δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα άρχεται. Πέρασε. Επίσης εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη J. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη L. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη M. Ποιο είναι υπέρ παρακαλώ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη T. Ταφ. Ε, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΑΕΦ. ΑΕΦ. ε, ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη AJ, ΑJ, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συνάδελφος Ροντ Α, όχι. Αιτιολογική σκέψη ΑΚ, ΑΚ. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το συνολικό κείμενο του ψηφίσματος ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Έκθεση ΒΟΟΝ για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Παράγραφος 5. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ε, Διανατάσεως. Παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 9 του αρχικού κειμένου. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το ε, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14 του αρχικού κειμένου κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 20 κατά τμήματα πρώτο τμήμα ονομαστική άρχεται πέρας Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ διανατάσσεω. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 25. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 26. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παραγράφος 34 κατά τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος παρακαλώ, διανατάσεως. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 60. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ Οκ. Θα ελέγξουμε την τροπολογία 5. Άρχεται λοιπόν ο έλεγχος της 5. Πέρας. Εγκρίνεται. Είχατε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ για την ε, συμβολή σας. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά άποχες. Να ελέγξουμε. Τροπολογία 2. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εντάξει. Εντάξει. Να ελέγξουμε και αυτήν. Είναι πολύ δύσκολο γιατί ένα 20% νομίζω ότι ψηφίζει. Ε, ε, ε προφορία, σε πάση περιπτώσει. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8, όπου έχει στηθεί ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9D. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Καλά, αν θέλετε να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται η ισοψηφία. Τροπολογία 10. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ωραία, αν θέλετε να ελέγξουμε και την 11. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 71. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Διανατάσεως παρακαλώ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά εντάξει, να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 ντε ονομαστική άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 ντε υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρασε. Απόρριτε. 15 υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχος. Καλός. Ε, πάντα το ίδιο συμβαίνει. Σας παρακαλώ ειλικρινά να σηκώνετε το χέρι σας. Το αποτέλεσμα πολύ συχνά ε, διαφέρει από αυτό που βλέπω. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 89 του αρχικού κειμένου ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε συνολικά το κείμενο υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Και συγχαίρουμε θερμά. Τον εισηγητή έκθεση Τσεσκόβα, τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Έχει καταπέσει οι 2. Α, θέλετε να ελέγξουμε την 1. Εντάξει, ωραία, ελέγχουμε την 1. Άρχεται. Πέρας. <clears throat> Εγκρίνεται. Οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Οπότε ψηφίζουμε, ε, τελείωσε η ψηφοφορία και θα περάσουμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου. Και σας εύχομαι καλή όρεξη.